Στη 14η Ιουνίου λοιπόν είναι μια σημαντική στιγμή και για την Εστονία και για όλη την Ευρώπη για τα κράτη αυτά τα οποία μπόρεσαν να ξαναβρούν την ανεξαρτησία τους. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει η συζήτηση για το θέμα αυτό και περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λάινεν για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Και θα δώσω πρώτα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Γεωλάινεν. Λάινεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα συζητούμε και αύριο θα ψηφίσουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα το οποίο εκ πρώτης όψεως δεν ίσως δημιουργεί μεγάλη εντύπωση, αλλά με το νομοθέτημα αυτό εμείς δημιουργούμε και ένα νέο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση Τη ευμάρειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε όλοι ότι το ΑΕΠ από καθαρά ποσοτική άποψη δεν επαρκεί για να απεικονίσει την ευμάρεια μιας χώρας, δεν λαμβάνει υπόψη την πτυχή την κοινωνική ούτε την πτυχή του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητο όμως εμείς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε έναν τρόπο να καταμετρούμε κατά πόσο εμείς προχωρούμε στα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε και υπέρ του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευμάρειας. Έχουμε τα στοιχεία της ε, αγοράς εργασίας. Έχουμε τα ετήσια στοιχεία για την οικονομία. Για τα θέματα αυτά έχουμε λοιπόν μία συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Αλλά όλα αυτά μας δίνουν απλώς ένα σκελετό και ένα είδος εμβαλωματικής εικόνας σε ό,τι αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος και μόνο. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε να έχουμε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των χωρών για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο απολογισμό για το κατά πόσο στα θέματα του περιβάλλοντος προχωρούμε προς τα εμπρός ή αν υπάρχουν πραγματικά υπαναχώρηση στα θέματα του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη το 2002 ζήτησε όλες οι πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με την κατάσταση του περιβάλλοντος να ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσον υπάρχουν τάσεις σημαντικές για τα θέματα αυτά και να υπάρξει και μια πληροφόρηση της κοινή γνώμης για τα θέματα αυτά. Και έχουμε καταλήξει σε έννοιες όπως είναι η χρήση των πρώτων υλών και του περιβάλλοντος για να μπορούν να ληφθούν υπόψη και από τους πολιτικούς λήπτες αποφάσεων. Τον Απρίλιο του 2010 η Κομισιόν λοιπόν προχώρησε με μια νομοθετική πρωτοβουλία και κατά την άποψή μας βέβαια δεν ήταν επαρκή αυτά τα οποία ξεκίνησε να κάνει η Κομισιόν. Είχαν ένα χαρακτήρα ο οποίος ήταν βραδιπορίας λιγάκι γιατί η Κομισιόν χρειάστηκε τόσο διάστημα για να αντιμετωπίσει ζητήματα τα οποία ήδη ο ΟΗΕ είχε αντιμετωπίσει πολύ νωρίτερα. Καταφέραμε λοιπόν να επιτύχουμε σημαντικέ προόδου με την δράση των πολιτικών ομάδων. Υπήρξαν δυσκολίε σε επίπεδο Συμβουλίου γιατί κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβαίνουν καθώς στην κατάρτιση των περιβαλλοντικών λογαριασμών, αλλά θα ήταν απαραίτητο να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση. Πρότεινε εδώ η Κομισιόν να υπάρξουν τρία επιμέρου στοιχεία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Καταρχήν οι εκπομπέ στην ατμόσφαιρα, που μπορούμε πολύ καλά να καταμετρήσουμε ποιες είναι οι εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα. Δεύτερον, οι χρηματοοικονομικές ε, ροές που έχουν να κάνουν με τους φόρους για το περιβάλλον και τις δαπάνες για το περιβάλλον. Και τρίτον, την ε, σχέση εισρωών και εκροών σε κάθε κοινωνία, οι ποσοτικές λοιπόν ροές σε σχέση με το περιβάλλον. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Ε, το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει ένας απολογισμός σε σχέση με τα, τους υδάτινους πόρους, με την ενέργεια, με τα απόβλητα και επίσης σε σχέση με την κατάσταση των δασών. Αυτά είναι τα βασικά συστατικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει βέβαια το επίμαχο σημείο το στατιστικό σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον για την αλληλεία, για τη θάλασσα κτλ. και την ρήπανση και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουμε κατορθώσει πιστεύω να καταλήξουμε σε κάποιες πρόοδους γιατί η Κομισιόν μέχρι το 2013 θα πρέπει να μας δώσει μια έκθεση για τα θέματα αυτά και να προβούμε ενδεχομένως σε μια αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Ελπίζω ότι μετά από την ε, διετία αυτή θα μπορούμε πραγματικά να μιλάμε για ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό ΑΕΠ και όχι μονάχα για το οικονομικό ΑΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, για την ε, παρουσίασή σας και για το γεγονός ότι τηρήσατε μέχρι κεραία στον χρόνο ομιλία σας. Ο κύριος ο Επίτροπος κ. Σόλυρεν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπε και ο εισηγητής ε, ε, Γιολάινεν, ο σκοπός της Επιτροπής και της προτάσεώς της ε, ήταν ακριβώς να υπάρξει κοινό νομοθετικό πλαίσιο για την συλλογή, συγκέντρωση και χρήση των ε, στοιχείων, των στατιστικών στοιχείων για τους οικονομικούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς ε, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη που όλοι επιθυμούμε. Με την παρουσίαση της προτάσεως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πρώτο στοιχείο του οδικού χάρτη πέρα από το ΑΕΠ στην Ευρώπη γίνεται μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και επομένως μέσω του τρόπου αυτού θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, τους οικονομικούς και τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς και όσοι λαμβάνουν αποφάσεις για την πολιτική θα διευκολυνθούν οπωσδήποτε. Ε, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των τριών θερμιστικών οργάνων και ακριβώς μέσω της συνεργασίας αυτής ε, επιτύχαμε την εφαρμογή αυτού του πλαισίου στην τηλεπικοινωνική πολιτική αυτό ε, περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία δηλαδή εκπομπές ε, ρήπων, ε, την ροή, τους λογαριασμούς ροής υλικών, καθώς επίσης και στοιχεία όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς φόρους που επιβάλλονται. Βεβαίως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε ε, να αποφευχθεί οποιοδήποτε επιπλέον βάρος των, ε, οργανισμών που θα πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία αυτά. Με τον κανονισμό αυτό ε, καθορίσαμε, δημιουργήσαμε μια πολύ ικανή βάση για, την, ε, ε, για τα στατιστικά δεδομένα και για τη διασύνδεση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας και πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει στο μέλλον όπως ακριβώς αναφέρεται και στην έκθεση. Ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ορίμανσης ε, ας πούμε ε, υλικά ξυλίας, αλληλεία κτλ. τα οποία θα μπορέσουν να ενσωματωθούν κάποια στιγμή. Οπωσδήποτε θα μας δίνεται σιγά σιγά η δυνατότητα να προσθέτουμε και άλλα modules τα οποία θα ενσωματώνονται σιγά σιγά στο κυρίως σώμα του πλαισίου αυτού αυτό που μας ενδιαφέρει και αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι κάθε τρία χρόνια θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση ε, των υπαρχόντων modules και ε, ενδεχομένως ε, να γίνεται προσθήκη καινούριων modules. Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι βουλευτές, επιτρέψτε μου τελειώνοντας να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Γιώ Λάινεν, ε, τον σκιώδη εισηγητή κύριο Μάρτιν, καθώς επίσης και όλα τα μέλη ε, των ε, Επιτροπών Περιβάλλοντος και Οικονομική, και η Οικονομική Επιτροπή για την πολύτιμη στήριξή τους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, εξ ονόματος όλων των βουλευτών. Ο συνάδελφος Μάρτιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν επανέλθουμε ε, στις πολιτικές θέσεις που είχε και ο κύριος Λάιν και εγώ την προηγούμενη δεκαετία είχαμε κοινέ θέσεις πολλές φορέ. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Είναι ουσιώδες, Είναι το πιο σημαντικό να μπορούμε να έχουμε στατιστικές οι οποίες είναι ελκυστικές, είναι σεξι. Μπορούν να μα δίνουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αξιοπιστίας που έχουμε εναντίον των ε, πολιτών. Γιατί πολλέ φορέ οι πολίτε θεωρούν ότι βλέπουν μονάχα τι λεπτομέρειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα ουσιαστικά θέματα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να μπορώ να μιλήσω σαν ανεξάρτητος βουλευτή, αλλά ω κάποιο ο οποίο είχε αντιμετωπίσει το νομοθέτημα αυτό ως σκιώδης εισηγητής και ως συντάξης γνωμοδότησης στην Επιτροπή Νομισματικών, Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Με 37-0 η Επιτροπή μας υποστήριξε αυτή τη θέση, κάτι το οποίο σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι θέλουμε να έχουμε πραγματικά στατιστικές για την αηφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μπορέσει να δώσει πραγματικά για τους νέους, για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ενιαίων στόχων και για το περιβάλλον και όχι απλώς να αποδίεται η Ευρώπη σε ένα ομό και βίαιο ανταγωνισμό με, την Ευρω... με ε, τις Πολιτείες, την Κίνα και την Ιαπωνία. Αυτό σημαίνει, όπως είπε και ο Γιώ ότι χρειαζόμαστε να έχουμε και πρόσθετα μότζους, πρόσθετα συστατικά στοιχεία. Υπάρχουν τέτοια ε, στοιχεία συστατικά τα οποία έχουν εκπονηθεί ήδη και στο παρελθόν. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να επιταχύνει τις ενέργειες της κατεύθυνση αυτή και θα ήταν χρήσιμο και από την πλευρά της Eurostat να υπάρξει μια μεγαλύτερη πρόοδος για τη συλλογή δεδομένων όταν έχουμε προβλήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα και η θέση μας ήταν σαφής 37-0 ότι πράγματι υποστηρίζουμε μια κίνηση της Κομισιόν προς την κατεύθυνση των στατιστικών του περιβάλλοντος με άλλα λόγια η Κομισιόν να χρησιμοποιήσει περισσότερους υλικούς πόρους και περισσότερους ανθρώπινους πόρους που έχουν προκύψει από τη διεύνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους θέσει στην υπηρεσία αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρήματο για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμού. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χώστα Σνέλχαρτ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Όταν διάβασα για πρώτη φορά την έκθεση της Κομισιόν ήμουν λιγάκι σκεπτική Είναι θετικό ότι υπάρχει κάποια κίνηση για τα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπανε οι προλαλήσαντες μου είναι ορθό ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα για τα θέματα αυτά. Στα περισσοτερα κάτι κράτη-μέλη υπάρχουν πάρα πολλά οικονομικά στοιχεία και στοιχεία τα οποία μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των διαφόρων modules, των διαφόρων τμήματων αυτού του απολογισμού και είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε σε όλες τις χώρες να έχουμε τις υλικέ ροές, τους φόρους του περιβάλλοντος και τις πηγές και την έκταση της ρήπανση στο περιβάλλον. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε σε πόσο εξαρτάται η οικονομία μας από το περιβάλλον αλλά και πώς θα εξασφαλίσουμε μια πιο αηφόρο πολιτική για το περιβάλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους μας. Τώρα, Μιλάμε πάντα για την ε, μείωση της γραφειοκρατίας κάθε φορά που βγάζουμε και ένα λόγο την Κυριακή ενώπιον των πολιτών. Και θέλω να επανέλθω και να πω προς την Κομισιόν είναι απαραίτητο να υπάρξει αυτή η μείωση της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν η πρότασή της είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στην Κομισιόν ή αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν και να μεταφέρουν προσωπικό το οποίο υπάρχει ήδη. Είναι απαραίτητο η συλλογή των στατιστικών στοιχείων που θέλουμε για το περιβάλλον να μην μας οδηγήσει σε περαιτέρω ε, επιβαρύνσει σε επίπεδο προσωπικού. Και όταν έχουμε την πρώτη έκθεση τη Κομισιόν το 2013, τότε θα πρέπει πραγματικά να πάρουμε και την απόφαση ποια είναι τα modules, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα χρειαστούν να προσθεθούν, γιατί μόνο τότε θα έχουμε μια κάποια εικόνα για το πώς έχει εξελιχθεί αυτό το σύστημα και να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία. Εγώ ένιωσα κάποιο τρόμο για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συζήτησε όλα αυτά τα θέματα ουσιαστικά γιατί έχουμε κάτι το οποίο είναι καινούριο και θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Η κυρία Ουλσκοκ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε μια πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε πραγματικά τι γίνεται στον τομέα του περιβάλλοντος και της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε καλύτερες δείκτες στη διάθεσή μας. Να μπορούμε να έχουμε τους ε, ενδείκτες οι οποίοι μας δείχνουν πώς εξελίσσονται οι συνθήκες στο περιβάλλον, στη βιομηχανική ανάπτυξη, αλλά και πώς συνδέονται τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε τις ορθές αποφάσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μεταλλαγές αν δεν έχουμε την πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία. Τώρα υπάρχει πια δυνατότητα να συλλέξουμε αυτά τα στοιχεία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε και μια σωστή απεικόνηση του ΑΕΠ ώστε να μην περιλαμβάνει μονάχα ε, οικονομικά στοιχεία, αλλά να έχει ένα διευρυμένο ορίζοντα. Είναι απαραίτητο επίση να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη συλλογή και τον συντονισμό των περιβαλλοντικών στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια καλύτερη λειτουργία των στατιστικών απεικονίσεων για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διαμόρφωσης με συντονισμένο τρόπο των πολιτικών περιβάλλοντα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην καταλήγουμε σε πολιτικές οι οποίες μπορεί να είναι και αντιπαραγωγικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αποφάσεις μας να εξασφαλίσουν για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δίδομαι προτεραιότητα στην ποιότητα η ποιότητα των πολιτικών και, των, και τις καλύτερες χρήσεις των πόρων και όχι μόνο μια πολιτική ποσοτική αντιμετώπιση. Ο κύριος Γιάντερ Μπράντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή κύριο Λάινεν για την έκθεσή του. Χρόνια ολόκληρα συζητάμε το θέμα αυτό και τώρα φαίνεται ότι επιτέλους προχωράμε με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το οικονομικό μας σύστημα αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και είναι απαράδεκτο αυτό το γεγονός και το κόστος που μεταφέρεται ολόκληρο στην κοινωνία. Γιατί να είναι πιο ακριβή η καθαρή ενέργεια από την συνήθη. Γιατί πρέπει πρώτα να καθαριστεί το περιβάλλον και τα έξοδα αυτά δεν τα πληρώνουν οι εταιρείε αλλά η κοινωνία. Δεν είναι λοιπόν μόνο τεχνική η έκθεση, είναι πολύ σημαντική γιατί η μέτρηση των πραγμάτων είναι γνώση τους όπως λέει μια Ολλανδική παροιμία. Έτσι λοιπόν στόχος είναι πώς θα καταλήξουμε σε μια πραγματικά βιώσιμη οικονομία. Θα ήθελα να δηλώσω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ότι για τα στοιχεία που έχουμε εδώ μπροστά μας πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση με βάση αυτά τα στοιχεία. Να δούμε δηλαδή αν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που εμπεριέχουν ή όχι. Θα ήταν λυπηρό αν δεν μπορούσαμε. Και ελπίζω από βάθος καρδίας να επιτρέψει η συλλογή όλων αυτών των στοιχείων να καταλήξουμε στην απομάκρυνση όλων αυτών των τοξικών και δηλητηριωδών ουσιών που συσσωρεύονται στο περιβάλλον. Ευχαριστώ πάντως ακόμη μια φορά τον εισηγητή. Είναι μια αρχή και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε για να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τη γνώση που διαθέτουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τρεμόπουλος από τους Πράσινους. Πρόεδρε, ευχαριστώ είναι δεδομένο και με όσα ακούσαμε μέχρι τώρα και από την έκθεση ότι χρειάζεται μια τεκμηριωμένη αξιολόγηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής ε, η οποία, η οποία χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα. Χρειαζόμαστε λοιπόν την ε, υποχρεωτική και εναρμονισμένη συλλογή τους. Όμως, οι συμβατικοί εθνικοί λογαριασμοί εστιάζουν κυρίως στις συναλλαγές της αγοράς και σε δείκτες που αντανακλούν σημαντικούς μεν παράγοντες στη δημιουργία ευημερίας αλλά δεν μετρούν την ίδια την ευημερία. ωστόσο υπάρχουν ε, οι νέες ελλείψεις φυσικών πόρων. Ε, χρειαζόμαστε άλλη όθηση στην παραγωγικότητα αλλά και ποιότητα. υπάρχει επιβάρυνση στους φυσικούς αποδέκτες με το να μην ε, δίνονται λογαριασμοί για το ιδιωτικό και το κοινωνικό κόστος της χρήσης των φυσικών πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος οι συμβατικοί λογαριασμοί μπορεί να στέλνουν λάθος μηνύματα προόδου στους φορείς λήψης των αποφάσεων οι οποίοι τότε μπορούν να βάλουν την κοινωνία σε έναν δρόμο μία αηφόρου ανάπτυξης. η εισαγωγή των περιβαλλοντικών και οικονομικών λογαριασμών έχει ουσιώδη σημασία αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσει την ανάπτυξη εναλλακτικών προς το αεπ δικτών οι οποίοι θα καλύπτουν τις διάφορες περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις. η επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις πριν από την έναρξη της περίοδου του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να θεσπιστεί μια περιορισμένη δέσμη σύνθετων δικτών που θα χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα του αεπ στη χάραξη της πολιτικής. σε αυτούς θα πρέπει να περιλαμβάνονται ένας νομισματοποιημένος δείκτης όπως οι προσαρμοσμένες καθαρές αποταμιεύσεις και ένας φυσικός δείκτης όπως το οικολογικό αποτύπωμα το αποτύπωμα άνθρακα ε, για την περιβαλλοντική διάσταση καθώς και κοινωνικοί δείκτες που ενσωματώνουν την κοινωνική διάσταση όπως μια εκτίμηση των ανισοτήτων όπως ο δείκτης τζίνι και ένας δείκτης κοινωνικής ένταξης και ανθρώπινης ευημερίας όπως ο δείκτης ανθρώπινης φτώχειας η αρχική πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει μόνο τη συγκέντρωση και συλλογή δεδομένων όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, τους περιβαλλοντικούς φόρους και επιβάλλονται στις διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, καθώς και τους μακροοικονομικούς λογαριασμούς για τη ροή υλικών. Έχουμε μια σειρά προτάσεις και τροπολογίες που κατατέθηκαν και πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη έκθεση αλλά και μια πρόοδο στο θέμα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, colleague. Ε, Ευχαριστώ. Να σας ζητήσω να μιλάτε με αργότερο ρυθμό. Είσαστε πάρα πολύ γρήγορος και η διερμηνία δυσκολεύεται να βγει στην ποιότητα που πρέπει. Paul Νούιταλ ε, Κύριε Πρόεδρε. Ε, για τους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λογαριασμού ακούγεται πάρα πολύ βαρετό πράγμα ε, και πίσω από αυτή την βαρεμάρα κρύβονται πολλά επικίνδυνα για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Α είμαστε ειλικρινεί. Ε, στην ουσία πρόκειται για εκπομπές, και εκπομπές ρήπων και περιβαλλοντικές φορολογίες. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει η Eurostat να δώσει περισσότερα στοιχεία. είμαστε πάλι ειλικρινεί. Ε, στην ουσία θέλετε περισσότερα στοιχεία έτσι ώστε να ελέγχετε περισσότερο και να φορολογείτε περισσότερο. Πέστε το καθαρά. Εν πάση περιπτώσει όμως το σημαντικότερο είναι ότι εδώ πρόκειται για κανονισμό όχι για οδηγία ε, και οι ε, κανονισμοί είναι αυτοί οι οποίοι ξεπερνούν ε, τον ευρωπαϊκό, τους εθνικούς νόμους και είναι αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν από την πίσω πόρτα να ξεπεράσουν και προβλήματα που δεν θα ξεπερνιόταν από το δικό μας κοινοβούλιο, από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μάρκιν, ο κ. και ο κ. Ε, Ζέπερ έχουν ζητήσει να χρησιμοποιήσουν την μπλε κάρτα. Όλοι μας είμαστε εδώ μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει και οι Βρετανοί να το κατανοήσουν αυτό. Δεν μπορούν, ελπίζω ότι μπορούν να μας δώσουν την απάντηση. Μιλήσαμε για την Σοβιε... Μιλήσατε για τη σοβιετοποίηση των στατιστικών. έτσι. Είναι η συλλογή στατιστικών στοιχείων σοβιετοποίηση, δεν θέλετε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση ευμάρειας, ε, την, ε, τον πληθωρισμό, την κατάσταση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Όλα αυτά δεν βοηθούν στον πολίτη να έχει μια καλύτερη εικόνα και δεν πρέπει οι λήπτες αποφάσεων και οι πολίτες να έχουν μια πρόσβαση σε καλύτερες και πιο αξιόπιστες στατιστικές. Ή όλα αυτά θα βλέπετε ότι είναι μια σοβιετοποίηση της Μεγάλης Βρετανίας. Ευχαριστώ, Λεωπρόεδρο. Να σας πω. Εδώ θέλετε πάντα να τα ελέγχετε όλα με συγκεντρωτικό τρόπο. Και σας λέω ότι οι επίτροποι δεν έχουν εκλεγεί από το λαό. Η δημοκρατία έχει σημασία για όλους. Ναι, πράγματι πιστεύω ότι βλέπουμε μια σοβιετοποίηση να δίνεται όλη η εξουσία στα Σοβιέτ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών. Το γεγονός ότι οι κανονισμοί μπορούν να παρακάψουν τα εθνικά κοινοβούλια, να παρακάψουν αυτούς που τους εξέλεξαν οι πολίτες Βρετανίας, είναι πραγματικά έσχος και είναι σοβιετοποίηση της Ευρώπης. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο Ρίχα Τζέμπερ έχει το λόγο. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Είχα ζητήσει και εγώ να θέσω ένα ερώτημα με μπλε κάρτα, κύριε Πρόεδρε. Ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Ο πρόεδρο χωρί μικρόφωνο. Αν μπορείτε να συνεχίσετε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημά μου. Η Μεγάλη Βρετανία όπως και άλλες πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει μια διαδικασία για την δημιουργία αυτών των λογαριασμών του περιβάλλοντος και όπως έδειξε και η θαυμάσια εργασία του Ιω είναι απαραίτητα αυτά τα στοιχεία, δεν έχει καμία σχέση με σοβιετοποίηση. Είναι στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να έχουμε μια συγκρισιμότητα βασικών στοιχείων πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε με τον τρόπο αυτό μια συγκεκριμένη συνολική λογιστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αφορά λοιπόν και την ε, Μεγάλη Βρετανία. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να έχουμε κοινά πρότυπα για να μπορούμε να καταμετρούμε την ευμάρεια και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών μας με συγκρίσιμα στοιχεία. Είναι κάτι που στο παρελθόν γινόταν με βάση το δολάριο. Είναι ευκαιρία να γίνεται τώρα και με βάση το ευρώ. Επίσης γνωρίζουμε ότι η κοινή αυτή μακροοικονομική αντιμετώπιση για όλη την Ευρώπη έχει πολλά ε, προβλήματα. Ξέρετε ότι η Φουκουσίμα θα παρουσιαστεί στο Ιαπωνικό ΑΕΠ σαν ένα θετικό αποτέλεσμα και θα οδηγήσει σε πολλές επενδύσεις. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ποιες είναι οι ροές και ποιες είναι και οι επιπτώσεις. Γι' αυτό τονίζουμε τη σημασία του να αναπτύξουμε μια νέα αντιμετώπιση για το ΑΕΠ που να λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό κάνουμε εμείς το πρώτο αυτό βήμα προς μια αηφόρο μορφή ΑΕΠ. Η ενέργεια παραγωγής χάρη, το να μπορούμε να έχουμε μια μικρότερη εξάρτηση από την ενέργεια μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στο ΑΕΠ, ενώ είναι θετικό για την ευμαρία μας. Γι' αυτό ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε στοιχεία τα οποία θα κάνουν την πολιτική μας πιο ελέγξιμη και πιο συγκρίσιμη. Τι κάνουμε με τις πρώτες ύλες, τι κάνουμε με τη ρήπανση. Αυτό θα βοηθήσει καλύτερα την ε, νομοθετική διαδικασία. Ακόμα και αν δεν ήσασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιείτε αντίστοιχε μεθόδου για να έχετε αξιόπιστα στοιχεία από τον οποίο να βασίζετε τι λήψει αποφάσεων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εμά και για την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Κρήτον Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα και με τη σειρά μου να συγχαρώ ε, τον ε, Γιώ για την εξαιρετική δουλειά σε αυτή την έκθεση. Πραγματικά είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε στους περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς δεν μπορούμε πλέον να βλέπουμε την οικονομία και το περιβάλλον ξεχωριστά. αυτή η διπλή κρίση που μας χτυπάει περιβαλλοντική και οικονομική δεν μας αφήνει τέτοια περιθώρια. οι παραλογισμοί του παρελθόντος πρέπει να σταματήσουν. Ε, ανέφερε και ο κύριος Ζίμπερ το παράδειγμα για τη Φουκοσίμα. Ένα άλλο πιο απλό καθημερινό παράδειγμα, οι πυρκαγιές μια πυρκαγιά η οποία καταστρέφει ένα δάσος την βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρει δηλαδή το καθαρό νερό τον καθαρό αέρα και ούτω καθεξής τη δυνατότητα το πλαίσιο για να παράγεται τροφή που καταστρέφει την πολιτική κληρονομιά ενός τόπου που καταστρέφει την αγροτική παραγωγή στο αεπ θα μετρηθεί θετικά γιατί θα γίνουν επενδύσεις για την αποκατάσταση. Κι όμως αυτή η χώρα, αυτή η περιφέρεια, αυτή η περιοχή θα έχει πληγεί μακροχρόνια. Μακροχρόνια θα είναι φτωχότερη από ό,τι ήταν πριν. Οι περιβαλλοντικοί και οικονομικοί λογαριασμοί που, οι οικονομικοί λογαριασμοί που σήμερα δεν είναι τέλειοι. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα βήμα προς ορθότερες πολιτικές που θα βασίζονται σε μια πιο πλήρη, πιο αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας. Είναι ένα βήμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε συνέπεια στι πολιτικέ μα θα μα επιτρέψει να πετύχουμε διεθνεί δεσμεύσει αλλά και το στόχο να πρασινίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρίκα Μάνερ. Ένα ολόκληρο λεπτό. <laughs> Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον Λάινεν για την σημαντικότατη εργασία του το κείμενο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, το είπανε και άλλοι συνάδελφοι. Διότι επιτέλους στην πολιτική μας θα μπορέσουμε να έχουμε δίκτες για το περιβάλλον, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα των εκπομπών στον αέρα και το θέμα των ε, οικολογικών φόρων. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να επιδείξουν ρεαλισμό. Ξέρουμε ότι είναι διαφορετική η κατάσταση στις διάφορες χώρες, ότι έχουν διαφορετικά στατιστικά συστήματα. Δεν πρέπει, δεν θέλουμε να αυξηθεί η γραφειοκρατία. Το είπε και ο Επίτροπος. Υπάρχει επίσης το θέμα των συνθετικών στοιχείων των συνιστοσών της πολιτικής του 20. Ένα λεπτό τώρα για τον συνάδελφο Ρώση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός ενσωματώνεται στο, πλαίσιο των, στο νομοθετικό πλαίσιο των ε, δικτών, των οικονομικών δικτών. Ε, οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικονομικοί λογαριασμοί θα πρέπει να αποτελούν στήριξη των αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικούς και οικονομικούς ε, παράγοντες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και έλεγχος αποτελεσματικός στις περιβαλλοντικές πολιτικές των κρατών μελών, αλλά με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επιπλέον γραφειοκρατία. Γι' αυτό εμείς θα ψηφίσουμε αποχή. Ε, Από την άλλη πλευρά αναφέρεται ο εισηγητής την πιθανότητα και το ενδεχόμενο να προσθεθούν επιπλέον modules ε, σιγά σιγά. Ε, αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η ρήτρα αναθεώρησης με τον τρόπο, με τρόπο ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν και οι μέθοδοι καταγραφής και συλλογής αλλά και οι μέθοδοι χρήσης των στοιχείων αυτών. Και αυτό βεβαίως σημαίνει περισσότερα χρήματα και περισσότερο άχθος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σοφία Κονή, επόμενη ομιλήτρια, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κατ' εμέ πολιτική είναι η προσπάθεια εξεύρεσης των καλύτερων δυνατών λύσεων ε, στα προβλήματα τα οποία ε, προκύπτουν. Πώς θα γίνει όμως αυτό εάν δεν γνωρίζουμε καλά και τα προβλήματα αλλά και τις ενδεχόμενες λύσεις. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο Έχω ερώτημα και δεν αφορά μονάχα την περιβαλλοντική πολιτική. Επομένως, είναι απαραίτητο όσοι λαμβάνουν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο είναι απαραίτητο λέγω να έχουν όσο γίνεται πιο εξαντλητικά και πλήρη στοιχεία πάνω στα οποία να βασιστούν. Αυτό είναι και το συμπέρασμα στο οποίο έφτασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2006 όταν πρότεινε στα κράτη-μέλη να διευρύνουν τους εθνικούς λογαριασμούς ε, λαμβάνοντας υπόψη τα κυρίαρχα στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης. Χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρωτοβουλία αυτή αυτή γιατί δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε περισσότερα και για, τους, ε, για τις εκπομπές ρήπων και για την επιβολή περιβαλλοντικών τάξη, φόρων κλπ. Όμως ε, στη διάρκεια της ψηφοφορίας αύριο θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα συλλεχθέντα ε, στοιχεία είναι αξιόπιστα και θα πρέπει επίσης να βεβαιωθούμε ότι αυτή η προσέγγιση θα αφορά όλες τις χώρες μέλη. Όντως, πώς μπορούν να καθοριστούν ευρωπαϊκές πολιτικές εάν δεν έχουμε στοιχεία για την κατάσταση κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις χώρες μέλη. Τέλος, θα ήθελα να στηρίξω δύο σημαντικές και ισχυρές ιδέες των οποίων υπεραμείνεται το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την διαδικασία ε, πράξεων ε, κατά εξουσιοδότηση που θα πρέπει να αναθεωρείται ως διαδικασία κάθε πέντε χρόνια. Γιατί κάθε πέντε χρόνια υπολογίζουμε ότι θα πρέπει να χρειαζόμαστε νέα στοιχεία Παρόλα αυτά όμως ε, ε, πρόκειται για ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κάριν Κάντενμπαχ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Ιολάινεν για μια ε, ρύθμιση η οποία έχει καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ χρόνο. Εμείς ήδη πριν εκλεγούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει να υπάρξει μια μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη βάση για να μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε όσο το δυνατόν να εκμεταλλευόμαστε τις στατιστικές που υπάρχουν σε πολλά κρατη κράτη-μέλη σε ένα ευρύτερο, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και την κρίση αξιοπιστίας που έχει πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά. Βλέπουμε πολλές φορές να υπάρχει μία πόλωση μεταξύ της οικονομίας και του περιβάλλοντος, ιδίως από τα μέσα ενημέρωσης. Και η συλλογή αυτών των στοιχείων θα μπορέσει να μας δώσουν μία καλύτερη και πιο εξισορροπημένη αντιμετώπιση για την επίπτωση της οικονομίας στο περιβάλλον και του περιβάλλοντος στην οικονομία και μπαλίν και να καταλάβουμε πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο στοιχεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς οι οποίοι πρέπει να λάβουν πολιτικές αποφάσεις για να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να βελτιώσουν μια γενικά γενικότερα την κατάσταση και όχι μονάχα να μιλάνε για θέσει εργασία ή για βελτίωση του περιβάλλοντο, αλλά έχουν μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Όπω είπε και ο Γιολάιν, θα έπρεπε να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ σαν μόνο με, μεσομέτρηση, να έχουμε ένα κοινωνικό και περιβαλλοντικό προϊόν που θα καταμετρά την πρόοδο. Σήμερα κάνουμε τα πρώτα βήματα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτή τη μεγαλύτερη αξιοπιστία για την Ευρώπη στα θέματα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής οικονομίας και της κοινή καταμέτρησης της πρόοδου προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. κύριε Κρίστα Κλάσια. δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Ένα, μια καλή στατιστική, μια καλή συλλογή στοιχείων, μια καλή αξιολόγηση όλων των στατιστικών στοιχείων, αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των στατιστικών στα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλήγουμε στι σωστέ αποφάσει για το μέλλον. Να έχουμε στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά συγκρίσιμα μεταξύ όλων των κρατών μελών, αυτό είναι ο στόχο μα. Το ερώτημα είναι βέβαια τι μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, ποιε θα πρέπει να είναι οι αποφάσει για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εξισορρόπηση τη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προτείνει να ακολουθηθεί μια σειρά στόχων, τα τρία βασικά modules για την αηφόρο ανάπτυξη. Η φορολογία του περιβάλλοντος, οι εκπομπές και οι υλικές ροές. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την φυτική παραγωγή. Παραγωγή χάρη τα θέματα των δημητριακών, των ελαιόδων σπόρων κτλ. που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξη όσο ο εισηγητή και ορισμένοι συνάδελφοι. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν είμαστε μονάχα σε επίπεδο ευχολογίου, αλλά και σε επίπεδο εφικτότητος στην, ε, στη δράση. Όχι μονάχα να έχουμε μια γραφειοκρατία που θα συλλέγει όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να έχουμε αξιοπιστία στα στοιχεία αυτά. Και τονίζω και πάλι εδώ πέρα να λάβουμε υπόψη τη σημασία τη φυτική παραγωγή σε ό,τι αφορά τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την παραγωγή ε, και την, την παραγωγή οξυγόνου και την κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακος από, τα, από τη φυτική παραγωγή και από τα φυτά γενικά είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε σχέση με το περιβάλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν και μία αντιμετώπιση αυτού του τομέα. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι συλλογές στοιχείων δεν θα πρέπει να γίνονται σε βάρος της ανεξαρτησίας των κρατών μελών και σε βάρος της δημιουργίας μιας πρόσθετης γραφειοκρατίας και βάρους προς τα κάτι μέλη. Κύριος ε, Ταβάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφός μας ο Λάινεν, έχει κάνει μια θαυμάσια έκθεση την οποία μας παρουσίασε. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για την οικονομία μας και για την κοινωνία μας και το περιβάλλον. Στο πάνελ ΣΤΟΑ που ε, αντιμετωπίζει ως μέλος αυτού του πάνελ που είναι σημαντικό και για την αντιμετώπιση της ε, φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος θεωρώ ότι αυτή η πρόταση κανονισμού είναι πάρα πολύ σημαντική για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη χρήση της χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης των δυνατήνων πόρων και των υπολείπων πόρων. Γιατί πράγματι για τα θέματα των υδατινών πόρων και για άλλους πόρους δεν έχουμε στοιχεία τα οποία να είναι αξιόπιστα ως μέλος και της Επιτροπής Γεωργίας θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε με ένα σαφή τρόπο ποιες είναι η, ποια είναι η αξία για την κοινωνία μας του περιβάλλοντος. Πώς μπορεί να καταμετρήσει κανείς την προσθέμενη αξία του περιβάλλοντος ώστε να καταλάβουμε και με ποιο τρόπο, παραδείγματο χάρη, οι γεωργοί κατά τη διάρκεια της αγροτικής παραγωγής μπορούν να δημιουργούν ένα δημόσιο, ένα κοινό αγαθό για όλους. Έχουμε τα λεγόμενα παραπροϊόντα τα οποία παράγονται από τη γεωργία, τα οποία όμως δεν λαμβάνει υπόψη ούτε η πολιτική ούτε η οικονομία. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια σταδιακή καλύτερη εικόνα για όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, Λεοπρόεδρος. Ο κύριος Ρούμπικ για ένα λεπτό έχει το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Ζουρουμπίχ. Αμικρόφωνος ο κύριος Ρούμπιχ. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Τώρα λειτουργεί αυτό το μικρόφωνο. Οι στατιστικές είναι κάτι που οδηγεί σε πολλές διαμφισβητήσεις και συζητήσεις πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη προστασία των δεδομένων από τη μία πλευρά, αλλά και την ανάγκη συγκρισιμότητα και διαφάνεια. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και να, να εξελίξουμε και μία διαδικασία δειγματοληψίας η οποία να είναι πράγματι αυτοματοποιημένη και να μας επιτρέπει να κάνουμε μια αξιολόγηση του πώς λειτουργούν οι διαδικασίες αυτές. Το να έχουμε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία θα μας διευκολύνει στο μέλλον να μπορούμε να παίρνουμε πιο εύκολα πολιτικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Βέρτμαν έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε μια κοινή λογιστική στην Ευρώπη για την οικονομία και το περιβάλλον θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα στοιχεία του περιβάλλοντος στις διάφορες πολιτικές και να τα κάνουμε πιο ορατά. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τα στοιχεία, τα στατιστικά τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται για να έχουμε καλύτερα στοιχεία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τις ε, προκλήσεις, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, τις απώλειες της βιοπικιλότητας, της μόλυσης του περιβάλλοντος, την εξάντληση των φυσικών πόρων. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε μονάχα αν έχουμε τα καλύτερα και τα πιο αξιόπιστα στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διατυπώσουμε καλύτερες προγνώσεις για τις μελλοντικές τάσεις, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική πολιτική αηφόρου χαρακτήρα και να εκμεταλλευτούμε την προσθέμενη αξία που θα μας δώσει. Η κυρία Σαβέλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον κύριο Λάινεν για την εξαιρετική αναφορά του. Πιστεύω κυρίες και κύριοι ότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε επίπεδο όπου σπάνια συναντάμε σύγκρουση πια μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Αντίθετα έχουμε εισέλθει σε μια φάση αλληλεπίδρασης. Οι Ευρωπαίοι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση. Η έκθεση αυτή θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του τι γίνεται με το περιβάλλον στην ευρώπη. τρία στοιχεία θα ήθελα να τονίσω το ένα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη ε, υποστηρίζω τη διαδικασία ανανέωσης των στοιχείων κάθε πέντε χρόνια και επίσης ότι θα πρέπει να έχουμε μια κοινή καταμέτρηση προόδου του οτιδήποτε κάνουμε για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Τζαβέλα. Τώρα το λόγο θα πάρει για ένα λεπτό ο κύριος Ομπερμάγερ. Παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν θέλουμε εμεί να διατηρήσουμε το περιβάλλον και για τις μελλοντικέ γενιές θα πρέπει να μην διαχωρίζουμε την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος από την οικονομική λογική. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μακροοικονομικές κοινέ αναλύσεις και για το περιβάλλον και για το, την οικονομία και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό τον απολογισμό με έναν τρόπο που είναι αξιόπιστος. Αλλά όταν τώρα ζητάει κεντρικά η ευρωπαϊκή στοιχεία για τα, από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ευαίσθητα θέματα όπως είναι η ατομική πολιτική, η πολιτική για τα γονιδιώματα και να αντιμετωπίσει τις σκανδαλώδεις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν σε πολλά επίπεδα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πιο αποτελεσματικό και αποφασιστικό τρόμο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της, ε, του περιβάλλοντος και της οικονομίας και το ρόλο ιδίως των μεγάλων συγκροτημάτων, ομίλων και λόμπι. Έχετε το λόγο, κύριε Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι βουλευτέ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ υπεύθυνη και επικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Ε, συμφωνούμε με την ε, πρόταση αυτή από ό,τι καταλαβαίνω ε, σε πολλά σημεία σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς και επίσης συμφωνούμε ότι τα στοιχεία αυτά θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη. Να απαντήσω σε κάποια σχόλια τα οποία έγιναν. Πρόκειται για τον πρώτο το κανονισμό ε, με τρία modules, με τρία συστατικά στοιχεία Ε, και ε, τα επόμενα modules ε, προετοιμάζονται και θα είναι έτοιμος ο νέος κανονισμός περί τα τέλη του 2012. Επίσης προβλέπεται και ένα, μια τρίτη ομάδα συστατικών στοιχείων. Επομένως πρόκειται για μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται διαρκώς πρέπει να πω όσον αφορά μια παρατήρηση που έγινε ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω διοικητικό και γραφειοκρατικό άκτος για τις επιχειρήσεις γιατί θα χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες δομές. Ε, πρέπει να πω μάλιστα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αυτό το οποίο ηγείται ε, της διαδικασίας συλλογής ε, περιβαλλοντικών στοιχείων Όσον αφορά τώρα τις ε, ε, στατιστικές και αυτά που είπαν οι κύριοι Λάινεν και Μάρτιν, ε, είναι ορθά. Δηλαδή έγιναν πολλές προσπάθειες βελτίωσης του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, Η πρώτη νομοθετική πρόταση που έκανε η παρούσα Επιτροπή τη 10 Φεβρουαρίου παρελθόντος έτους ε, μετά την ε, θετική ψήφο ε, που δώσατε για την σύσταση της νέας Επιτροπής ψήφισε λοιπόν ε, μία ε, πρόταση για την Eurostat. Νέες δυνατότητες λοιπόν εδόθησαν στην Eurostat έτσι ώστε να ελέγχει στην πηγή την ορθότητα των στατιστικών στοιχείων. Uh, Δεύτερον, το σχέδιο δράσης για την ε, Ελλάδα εφαρμόζεται και μέσα σε ένα χρόνο οδήγησε ε, σε ε, εκβαθέων τροποποίηση του ελληνικού στατιστικού ε, συστήματος και είναι γεγονός επίσης ότι και όσον αφορά το υπερβολικό χρέος και αυτό έχει αρχίσει να μειώνεται. Τέλος, για τους πόρους. Δεν χρειαζόμαστε πόρους για αυτό το συγκεκριμένο θέμα των περιβαλλοντικο-οικονομικών λογαριασμών. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Μάρτιν ότι χρειαζόμαστε αρκετούς πόρους βεβαίως και... Θα συναντηθώ την επόμενη εβδομάδα ε, στο Λουξεμβούργο με τους επικεφαλείς της ε, Eurostat έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα των ε, πόρων και ε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε με νέο αποτελεσματικότερο τρόπο ε, τις, ε, τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας έτσι ώστε το αποτέλεσμα είναι πιο ικανοποιητικό. Πάντως ε, δεν μπορούμε να πάρουμε πόρους ε, από την διεύρυνση όπως ε, πρότεινε ο κύριος Μάρτιν γιατί είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για μας η πορεία προς την Ευρώπη των Δυτικών Βαλκανίων και επομένως δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο με ήπια δύναμη και με διαδικασία ε, διεύρυνσης θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις ε, χώρες αυτές. Αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, τώρα ο συγητής, ο κύριος Λένεν, έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. <coughs> Κύριε Συγητά. Yeah. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συζήτηση και για την ευρεία υποστήριξη που δείξατε για την δημιουργία των περιβαλλοντικών λογαριασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ελάχιστες ε, εξαιρέσεις υπήρξε υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή και μπορώ να συμμεριστώ και αυτά που είπε η κυρία Κάλεμπαχ. Πολλοί από εμά θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε αυτά να είχαν γίνει ήδη στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία διαθέσιμα και <clears throat> γι' αυτό είναι <clears throat> χρήσιμο να προχωρήσουμε για την κατεύθυνση αυτή. Όπως είπε και ένα συνάδελφος, το να μετράμε σημαίνει να γνωρίζουμε η βάση για όλη τη λήψη αποφάσεων και για όλα τα προγράμματά μας θα πρέπει να είναι η καλύτερη γνώση ώστε να είναι τεκμηριωμένες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε και επομένως αυτά, αυτή η οι ισολογισμοί του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντικοί και σας υπενθυμίζω και τον κύριο στόχο της στρατηγικής του, της Ευρώπης του 2020 η βιωσιμότητα και η αηφορία είναι πάρα πολύ σημαντική Εάν θέλουμε λοιπόν να είναι επιτυχής αυτή η στατιστική, θα πρέπει να έχουμε τρόπους μέτρησης της πρόοδου και ξέρουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώσουμε την καταμέτρηση του ΑΕΠ με μία μορφή απολογισμού για την φύση, για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους και για όλη την προβληματική της βιωσιμότητας. Κυρία Κλάσο, όλα αυτά λοιπόν δεν είναι υπερβολικό άχθος για τα κράτη-μέλη. Θα προχωρήσουν σταδιακά τα modules, όπως είπε και, ο, και η Επιτροπή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ήδη έχουμε από την νομοθεσία, πραγματικά για τα απορρίμματα, για τη ρήπανση, όλα αυτά τα στοιχεία να τα εκμεταλλευτούμε περισσότερο. Η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να λάβει υπόψη και την ανάγκη σε, δημο... σε όπως είναι αυτή για τη βιοποικιλότητα και για την κλιματική αλλαγή, να ξέρουμε σε ποια θέση βρισκόμαστε αν προχωρούμε ή δεν προχωρούμε στα θέματα αυτά. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν του σκιώδει εισηγητέ, θέλω να ευχαριστήσω και την Eurostat για το έργο το οποίο φέρνουν σε πέρα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στο Λουξεμβούργο, στη Eurostat, να καταρτήσουμε αυτού του ισολογισμού που να περιλαμβάνουν και το περιβάλλον. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τονίζω και πάλι ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα. Το αναγνώρισαν πολύ, ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε στο σημείο αυτό και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση της